8.000 νέοι και νεαροί άνδρες σε λίγες μέρες συστηματικά με συστηματικό τρόπο και κτηνόδη τρόπο δολοφονήθηκαν στην καρδιά της Ευρώπης αυτό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου στη Σρεμβρενίτσα συνέβη το χειρότερο έγκλημα πολέμου στην Ευρώπη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μια πραγματική πράξη γενοκτονίας που ποτέ δεν θα έπρεπε να είχε λάβει χώρα. Μια συλλογική αποτυχία της διεθνούς κοινότητας που μέχρι σήμερα μας έχει τραυματίσει και μας απασχολεί βαθύτατα. Γονατίζουμε μπροστά στα θύματα. Εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζω στους οικείους της οικογένειές τους και τους συγγενείς τους τα βαθύτερα, βαθύτατα συλληπιτήριά μας. Μέχρι τη σημερινή μέρα δεν έμαθαν όλοι, δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη σε όλους. Όσον αφορά όλους τους δολοφονημένους δεν βρήκαν τάφο όλοι. Και γι' αυτό πρέπει πραγματικά <clears throat> να δοθεί μάχη να δικαιωθούν οι οικοί και οι συγγενείς των θυμάτων όπως τους αξίζει το 2007 η γενοκτονία αυτή από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επιτέλους αναγνωρίστηκε ως γενοκτονία. Ήταν ένα σημαντικό ορόσημο αυτή η στιγμή τότε. Ιδιαίτερα επειδή η γενοκτονία συνέβη σε μια περιοχή που το ασφαλής από τα Ηνωμένα Έθνη τότε. Και αυτό ήταν, έγινε σύμβολο της διεθνούς κοινότητας που δεδομένων των σοβαρότατων παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου έγινε σύμβολο η Σρεβρενίτσα. Έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο φορές ήδη τοποθετηθεί το 2005 και το 2009 σε, στις δολοφονίες της Σρεβρενίτσα. Όλα τα θύματα τότε έτυχαν φόρου τιμής στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Απόψε 20 χρόνια μετά ανανεώνουμε αυτή τη δέσμευσή μας Τη Σρεμπρενίτσα δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Διότι η συμφιλίωση, κυρίες και κύριοι, χωρίς μνήμη δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση χωρίς μνήμη. Συμφιλίωση μπορεί να υπάρξει μόνο τότε όταν τα πάθη και τα δεινά του παρελθόντος τα αναγνωρίζουμε και όταν θυμόμαστε πώς ε, οι δηλητηριασμένοι λόγοι και το εθνοτικό μίσος τότε είχαν πάρει το πάνω χέρι όταν θυμόμαστε πόση πολυεθνοτική και πολύπλευρη ε, πολιτιστική και εθνοτική παράδοση στα Βαλκάνια ήταν κάτι το οποίο είχαν αρνηθεί κάποιοι και θέλησαν να καταστρέψουν βρισκόμαστε μπροστά σε όλους εκείνους που θέλουν να αναζωογονήσουν τα παλαιά δαιμόνια και θέλουμε να τους σταματήσουμε. Και γι' αυτό κυρίες και κύριοι τέτοιου είδους φόροι τιμής είναι σημαντικές εκδηλώσεις ώστε να συνειδητοποιούμε κάθε φορά ποιες είναι οι καταστροφικές δυνάμεις εκείνες οι οποίες παραμένουν ακόμα ζωντανές στην, την συνάδελφο κυρία Αντιπρόεδρο Λούνατσεκ παρακάλεσα την επόμενη εβδομάδα να εκπροσωπήσει την ε, ενδεκάτη του μήνα στη Σρεμπρενίτσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άοκνα καταβάλει προσπάθειες για την ευρωπαϊκή προοπτική των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων και για μια σταθερή και ασφαλή γειτονική σχέση σε αυτή την περιοχή που είναι προς το συμφέρον μας. Η θύρα της Ευρώπης είναι ανοιχτή σε όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν την οδό της δημοκρατίας και τη συμφιλίωση. Η συμφιλίωση ως κλειδί για την ασφάλεια, συνεργασία και ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι να εγερθούμε και να αποτίσουμε φόρο τιμή στα θύματα της Σρεμπρενίτσα Σας ευχαριστώ. So, meine Damen λοιπόν,